πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως Ιταλοί, Εστονή και Βρετανοί υπήκοοι, οι οποίοι κρατούνται στην Ινδία. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στους συντάκτες των ψηφισμάτων. Πρώτος είναι ο κύριος Τάραντ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα ψηφίσματα αυτά Τα ψηφίσματα αυτά έχουν υποστηριχθεί από όλες τις πολιτικές ομάδες. Ερχόμαστε με κάποια καθυστέρηση, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα βοηθήσει να υπάρξει τέλος αυτή τη συζήτηση. Έχουμε το θέμα των ε, Ιταλών ναυτικών και επίσης πολιτών της Εστονίας και των, του Ηνωμένου Βασιλείου. Νομίζω ότι όλα αυτά δημιουργούν ακόμα πρόσθετα προβλήματα. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που οι Εστονοί βουλευτέ σε όλε τι πολιτικέ ομάδε έχουν αναγνωρίσει τη σημασία αυτού του προβλήματο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Καστάλτο, τον Μαντσέρη και την Κόμη από την Ιταλική Αντιπροσωπεία που κατάλαβαν πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό και τα έλαβαν όλα αυτά υπόψη του. Εγώ ελπίζω <clears throat> ότι θα μπορέσουμε με την κοινή αυτή υποστήριξη να θέσουμε το θέμα αυτό το οποίο συνδυάζεται με το θέμα των Ιταλών ναυτικών και θέλω να, ευχαριστήσω όλους αυτούς που με την έρευνά τους βοήθησαν για το ψήφισμα αυτό και πήραν πληροφορίες από την Ινδία. Έχουμε αυτό το κοινό ψήφισμα, θέλουμε να το παρουσιάσουμε. Δεν αναφέρουμε βέβαια την ειδική κατάσταση των Ινδικών δικαστηρίων. Δεν είμαστε διπλωμάτες, δεν εργαζόμαστε για διπλωματικές υπηρεσίες το ψήφισμά μας θα πρέπει να αντανακλά τα γεγονότα και την πραγματικότητα, αλλιώς δεν θα έχει το σωστό αντίκτυπο. <clears throat> Σε ό,τι αφορά το άρθρο 2 του κοινού ψηφίσματος, η Ινδία έχει πάνω από ένα δισεκατομμύριο κατοίκους, η Εστονία έχει λίγο παραπάνω από ένα εκατομμύριο. Περί μεγέθους ουδής λόγος. Επομένως, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπάρχει μια διαφορά σε ειδικό βάρος. Το ψήφισμά μας είναι ένα καλό ψήφισμα το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων αυτών και πιστεύουμε ότι και οι Βρετανοί και οι Εστονοί είναι άτομα τα οποία έχουν δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μποργέζο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω και την ομάδα μου που υποστήριξε σήμερα στην Ολομέλεια ένα ψήφισμα που σκοπό έχει να θίξει ένα σημαντικότατο θέμα για τη χώρα μας, την ε, Ιταλία. Δύο Ιταλούς ναύτες, εκ των οποίων ένας είναι ακόμη φυλακισμένος στην Ινδία, ο άλλος πρόκειται να δικαστεί. Εδώ ήταν τελείως αυθαίρετη η εκδίκαση των υποθέσεων και η όλη υπόθεση δεν φαίνεται να έχει λύσει θα ξεπεράσει και το 2018. Η Ιταλία είναι μια μεγάλη χώρα, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεγάλη όμως ε, χώρα πρέπει να υπερασπίζεται και τους πολίτες της και που είναι φυλακισμένοι στο εξωτερικό. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να λέμε αντικειμενικώ ότι έγιναν πολλά με τόσο ισχνή υπεράσπιση και πολλές φορές με ε, με κατασκευασμένα επιχειρήματα. Αυτό που γίνεται είναι ότι αποδυναμώνεται η υπεράσπιση των ε, κατηγορουμένων και στο ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να αναρωτηθούμε πού πήγε αυτή η Ευρώπη, δεν πρέπει να μας ε, υπερασπιστεί από το Ισλαμικό κράτος. Δεν μπορεί καν να υπερασπιστεί δύο στρατιώτες, οι οποίοι ούτως ή άλλως ε, είχαν επιδοθεί σε έναν αγώνα που μας αφορά όλους, την τιμωρία της διεθνούς πειρατείας θα έλεγα ότι πρέπει και ένα άλλο σημείο να προσπιστούμε, δηλαδή των στρατιωτών μας, της στρατιωτικής τιμής. Αυτό διακυβεύεται εδώ και αυτό ίσως να είναι και ο λόγος της ε, ισχνής αυτής ε, προσπάθειας για να προσπιστούμε αυτούς τους πολίτες. Δεν φαίνεται η προσωπική ασφάλεια των πολιτών της Ένωσης να αφορά τα θεσμικά όργανα. Για, ένα τέτοιο, για μια τέτοια σκοτεινή υπόθεση που τόσο αργά πήρε την κατεύθυνση της ε, διεθνούς επίλυσής της. Η ευρωπαϊκή φωνή πρέπει να υψωθεί γιατί πέραν της είπα της εκπροσώπου Μογκερίνη είδαμε να μην υπάρχουν ε, αποτελεσματικές δράσεις. Θα έπρεπε όπως ναύτες μας που προασπίζονται τη θεμελιωτή ελευθερία στις θάλασσες και εμείς να προσπιστούμε τη δική τους. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει στο σύνολό της τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας ξεκινώντας από την αναστολή οποιοδήποτε διαπραγμάτευσης βρίσκεται σε εξέλιξη οποιασδήποτε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Ζήτω το στρατιωτικό ναυτικό στη Μεσόγειο και ζήτω το ιταλικό ναυτικό. Ελευθερία στους Ιταλούς ναύτες. Ευχαριστούμε κύριε Μποργέτζιο, η κυρία Αντινόλφη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι εδώ ο συντάκτης του ψηφίσματος και δεν μπόρεσε να ε, παραστεί για τη συζήτηση. Το Κοινοβούλιο καλείται να εκφραστεί για μια περίπτωση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων για άλλη μια φορά. Είναι η περίπτωση της σύλληψης και της καταδίκης 35 υπηκών από τη Βρετανία και την Εστονία και όπως υπόθηκε προηγουμένως και δύο Ιταλών ναυτών. Ε, υπ' αυτήν την έννοια, ε, ε, καθήκον μας είναι τα κράτη-μέλη σήμερα να δείξουν την ίδια συνοχή όπως και στο παρελθόν. Χρειάζεται συντονισμένη δράση από την πλευρά ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας στην πραγματικότητα και θα είχαμε προλάβει ήδη να δώσουμε μια ικανοποιητική λύση στην όλη υπόθεση. Γι' αυτό η ύπατη πρόσωπος, η κυρία Μογκερίνη, θα έπρεπε να έχει αναλάβει δράση πολύ νωρίτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φανόρντεν. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της ε, πειρατείας απεδείχθηκε ότι είναι η χρήση ομάδων ασφάλειας ε, ε, που επιβαίνουν στα σκάφη ε, συγκεκριμένα στα μετρικά σκάφη που ουσιαστικά είναι σαν ε, πλωτά όπλοστάσια ε, και προστατεύουν τα σκάφη που χρήζουν προστασίας. Αυτό του είδους λοιπόν το πλωτό οπλοστάσιο ήταν και το σκάφος MV Seaman Guard Ohio. το οποίο το στις 12 Ιανουαρίου συνελήφθη το πλήρωμά του ε, στην πολιτεία Ταμίλ Ναντού. 35 άτομα κρατούνται. Υπάρχουν κάποια νομικά επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Ε, δυστυχώς ε, με βάση αυτά τα επιχειρήματα καταδικάστηκαν και σε πενταετή κάθεξη που είναι η υψηλότερη ποινή. Και παραμένουν αυτή τη στιγμή σε κράτηση στην Ινδία. Φυσικά και έχει αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει και κυριαρχία, ε, γνωρίζουμε την παράδοση της χώρας, γνωρίζουμε ότι έχει πληγεί από, από τρόπες τρομοκρατικές ε, επιθέσεις η χώρα που πολλές φορές διενεργούνταν από θαλάσσεις. Παρ' όλα αυτά, ε, το προσωπικό αυτό, το πλήρωμα αυτού του πλοίου ούτε επικίνδυνο ήταν, ούτε άσκησε βία, ε, ούτε είχε κάποια δράση κατά των συμφερών της χώρας. Αντιθέτως ε, δρούσε προστατεύοντας, καταπολεμώντας την πειρατεία. Οι Ιστανοί, οι Εστονοί, οι Βρετανοί ναυτικοί είναι η τύχη τους άγνωστοι, νιούν τα μέλη των οικογενειών τους. Πρέπει να τηρηθούν ιδέωσες διαδικασίες και θα πρέπει να λήξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το θέμα θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος, ε, από τον κύριο Ντέβα, παρακαλώ, έχετε μια γαλάζια κάρτα, τη δέχεστε. Κύριε Ντέβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Φίλος μου, ο κύριος Βαν Όρντεν, δέχεται ότι είναι παράλογο οι ειδικέ αρχές να έχουν ε, την ίδια αντιμετώπιση για όλους ε, που καταδίκασαν αυτούς τους ανθρώπους. το πλήρωμα έπρεπε να υπακούσει. Και αν δεν είχε υπακούσει θα τους είχαν ε, για ανταρσία ε, εκτελέσει. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν καταλαβαίνουν ε, οι Ινδικές Αρχές τι σημαίνει για ένα πλήρωμα να υπακούσει εντολές ή να μην υπακούει. Κύριε Ντέβαλε, κύριε Σανόρντ, είναι πολύ σωστό το επιχείρημά σας. Αδιάκριτες συλλήψεις και προσαγωγές ε, οι άνθρωποι αυτοί δεν κάναν και τίποτα ουσιαστικά οι ίδιοι, το οποίο να ήταν ε, παραπτωματική συμπεριφορά. Και πραγματικά, όπως είπε πολύ σωστά ο φίλος, ε, δεν μπορούσαν να δράσουν διαφορετικά. Γι' αυτό και ζητάμε να λήξει ώστε να το πιο γρήγορα αυτό το ζήτημα. Ο κύριος Κέλαμ έχει το λόγο ο συντάκτης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φανό Όρντεν για την εξισορροπημένη παρέμβασή του και για τη βοήθειά του στην προετοιμασία αυτού του εγγράφου. Δεν ήταν εύκολο, ήταν πολύπλοκο, αλλά φτάσαμε ένα σημείο όπου ήταν έτοιμο το ψήφισμα. Θέλω να εκφράσω επίσης την κατανόησή μου για τους δύο Ιταλούς ναυτικούς που βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση. Όλοι οι περισσότεροι από τους Ιταλούς ε, συναδέλφους μας τόνισαν ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να αποχωριστεί από τη σημερινή συζήτηση. Παρ' όλα αυτά εκφράζουμε την κατανόηση, τη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας προς τους Ιταλούς ναυτικούς. Αλλά εδώ πρόκειται για το μέλλον 20 πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 14 Εστονών και 6 Βρετανών οι οποίοι ασκούσαν αντιπειρατικές δράσεις κατά και των οποίων το πλοίο συνελήφθη από τους Ινδούς το 2013 μάλιστα. Αυτό που είναι το ενδιαφέρον είναι ότι δεν κατηγορήθηκαν για λαθρεμπόριο, για ένοπλη επίθεση ή οτιδήποτε τέτοιο. Απλώς κατηγορούνται για το γεγονός ότι μπήκαν στα χωρικά ύδατα της ε, Ινδίας ε, έχοντας όπλα. Και επειδή αγόρασαν ε, καύσιμα από μη επίσημες πλευρές. Νομίζω ότι θα είναι απαράδεκτο να θεωρήσουμε ότι μια τέτοια ε, διαδικασία αντί να κρατήσει κάποιους μήνες έχει κρατήσει πάνω από δύο χρόνια. Έχουν αθωωθεί από ένα ειδικό δικαστήριο αλλά έχουν καταδικαστεί από ένα άλλο πέντε χρόνια στη φυλακή. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να διαφυσβητήσουμε την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος της Ινδίας. Αλλά είναι μέσα στα πλαίσια ενός κλίματος φιλίας και αμοιβαίας κατανόησης είναι απαραίτητο να απελευθερωθούν αυτοί οι 20 άνδρες οι οποίοι έχουν ήδη φυλακιστεί για πάνω από δύο χρόνια. <clears throat> και είναι απαραίτητο να αγωνιστούμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο ιερό καθήκον των μελών του Κοινοβουλίου να ασχοληθούμε με το μέλλον των συμπατριωτών μας. Αυτό δεν μπορεί λοιπόν να εξαρτάται από διπλωματικά χρονοδιαγράμματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος. Ο κύριος Πάετ έχει το λόγο. Δεκατέσσερις Εστονοί και έξι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν εμπλακεί σε μια ατυχή κατάσταση στην Ινδία για πάνω από δύο χρόνια. Ενώ αθώθηκαν από όλε τι κατηγορίες το 2014, στο δευτεροβάθμιο επίπεδο την προηγούμενη εβδομάδα καταδικάστηκαν από το εφετείο σε πέντε χρόνια ε, φυλάκισης που ήδη εκτίουν. Αυτό μας σοκάρισε όλους. Ο στόχο του ψηφίσματο είναι να επιστήσουμε την προσοχή τη Ινδία αλλά και τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα αυτό, ώστε να μπορεί να προέλθει μια θετική λύση σε αυτό το πρόβλημα. Καταλαβαίνουμε τι ανησυχίε τη Ινδία και τι ευαισθησίε του. Ζητούμε να καταλάβει και τη δική μα άποψη. Οι άνδρες αυτοί ήταν σε αντιτρομοκρατικά καθήκοντα ω <coughs> ομάδα προστασία, που είναι το μόνο αποτελεσματικό μέτρο κατά των πειρατών. Γι' αυτό το λόγο χάνουν την ε, ελευθερία του και βρίσκονται μακριά από τι οικογένειε του. Θα πρέπει η Ινδία να μα βοηθήσει να του ξαναφέρουμε στα σπίτια του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Πιέρ Αντώνη Παντσέρη. Πρώτα πρώτα πρόεδρε, ήθελα να επισημάνω την ε, γραφειοκρατική δισκαμψία της Προεδρία διότι υπάρχουν αμφισημίες και σφάλματα που είναι πολύ ενοχλητικά στον τίτλο του ψηφίσματος αναφέρονται Ιταλοί αλλά τελικά δεν αναφέρεται καθόλου στο κείμενο, στο σώμα του ψηφίσματος το θέμα των Ιταλών ε, διαγράφηκε η παράγραφος αυτή θα έπρεπε λοιπόν να αλλάξει και ο τίτλος εφόσον κάνουμε αυτή τη συζήτηση διότι από ό,τι φαίνεται η επικοινωνία μας δεν ήταν αποτελεσματική σήμερα μιλάμε απλώς για, τους, ε, για τα μέλη της περιπόλου του Seaman Guard ε, Ohio που ήταν Εστονοί και Βρετανοί στο μεγαλύτερο μέρος τους. το ψήφισμα αυτό δεν είναι μια έκφραση καταδίκης της Ινδίας, μια χώρα που σεβόμαστε και που έχει δημοκρατική παράδοση. Απλώς έχουμε την απέτηση, μετά βλέπουμε, βλέποντας την ε, αμφισημία και την ολιγορία των δικαστικών διαδικασιών, ότι θα έπρεπε να εκδικαστούν οι υποθέσεις αυτές με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας μπορούν να βρεθούν θετικές λύσεις στην όλη υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Και τώρα για τις πολιτικές ομάδες από το ΕΛΚ ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι πεπισμένος με όλες τις πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οι πολίτες μάλλον και οι ναύτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελούσαν καμιά μορφή κίνδυνο για την Ινδία ούτε κάποιο είδου απειλή. Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να έχει επιληθεί πολύ νωρίτερα και η υπόθεση να έχει οδηγήσει σε μια δίκαιη λύση. Είναι απαράδεκτο όσο συμβαίνουν και υπάρχει μια αντίφαση στο πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται τα πράγματα και αντιδρά. Θα έπρεπε να δούμε ότι μεταξύ του 2010 και 2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση επέτρεψε στην Ινδία με ένα κοινό πρόγραμμα αξίας 470 εκατομμυρίων ευρώ ε, για τον τομέα της υγείας και άλλους τομείς διατέθηκαν στην Ινδία. Θα έπρεπε ενδεχομένως να επαναξετάσουμε την στάση μας αυτή. Ίσως δεν θα έπρεπε υλικά να στηρίζουμε καθεστώτα που ε, αντιμετωπίζουν κατά αυτόν τον τρόπο τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι πονίδιστη αυτή η συμπεριφορά. Με ευχαριστούμε. Εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Μαριού Λάουριστην. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι ιδιαίτερω που όλες πολιτικές ομάδες ομόφωνα σήμερα αποφάσισαν να, να δείξουν αλληλεγγύη προς ε, όλους αυτούς τους ναυτικούς των οποίων ε, η μοίρα ανησυχεί όλο τον ιστορικό λαό. Και βέβαια δεν μας απασχολεί μόνο το τι θα γίνει με τους εστονούς ναυτικούς, αλλά και τους Βρετανούς και τους Ιταλούς ναυτικούς. Μιλάμε για αλληλεγγύη προς τα έθνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για πολλά άλλα μεγάλα πράγματα όμως είναι και θέμα που αφορά την καθημερινότητα και αφορά και τον κάθε μεμονωμένο συνάνθρωπό μας η αλληλεγγύη. Κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μπορεί να πιστεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεματοφύλακα υπέρμαχο της αλληλεγγύης και αυτή είναι η συμβολική αξία αυτού του ψηφίσματος. Όλοι οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι είναι ίσοι και ε, αξίζουν τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κύριο Ντέβερ τώρα το λόγο. Το ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω πρόβλημα που γίνεται αυτή η συζήτηση, αλλά το έχω ξαναπεί. Ρωτώντας τον κύριο Βαν Όρντεν μετά την ομιλία του ότι δεν μιλάμε μόνο για το δικαστικό ατόπιμο εδώ, αλλά και πώς θα βοηθήσουμε τους Ινδούς να εξυγχρονίσουν το δικαστικό του σύστημα. Διότι για τους ανθρώπους αυτούς που συνελήφθησαν. Επί δύο χρόνια ε, ήταν σαν αστολή. Δεν υπήρχε καμία δυνατότητα να κάνουν κάτι περισσότερο. Δύο χρόνια χρειάστηκε να, δικαστεί, εκδικαστεί η υπόθεση. Υπάρχουν ε, μέχρι και 20 χρόνια ε, αναμονή για τις δίκες. Ε, καταραίει το σύστημα. Αν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε την Ινδία. Αυτό είναι να βοηθήσουμε να εξυγχρονίσει τις νομικές δικαστικές της δομές. Thank you. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους της Άλντε. Κύριε Γιάννα Τόμ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φύλακες του εσθονικού πλοίου καταδεικνύουν ότι όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να αντιμετωπίσουν αντιστοιχά προβλήματα. Η Ινδία είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε όμω ότι η ύπαρξη δημοκρατικών διαδικασιών δεν σημαίνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, εξασφαλίζονται και υπάρχει το δικαίωμα για δίκαια δίκη. Δεν θέλω τώρα να αξιολογήσω τα ειδικά δικαστήρια ή την ειδική δικονομία, αλλά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αυτή η διαδικασία <clears throat> κράτησε πάρα πολύ χρόνο. Η Εστονία και οι Εσθονοί και άλλοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν βρεθεί σε μια πολύπλοκη κατάσταση. Οι φύλακες των πλοίων έχουν χρειαστεί να δανειστούν για να διαθρέψουν την οικογένειά τους αυτά τα δύο μισή χρόνια γιατί δεν μπορούσαν να εργαστούν και τα προξενία της Εστονίας και της, ε, της Εστονίας ε, είναι με πολύ περιορισμένη σύνθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν όλα αυτά που είναι δυνατά ώστε να δώσουμε διπλωματική βοήθεια σε όλους. Από την ομάδα EFTT ο κύριος Άρνοτ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Έχω κάθε σεβασμό για τον ειδικό λαό και την ειδική κυβέρνηση. Σέβομαι την κυριαρχικότητα της χώρας αυτής και αναγνωρίζω τις δυσκολίες που προκύπτουν σε μια παράδοξη κατάσταση η οποία δεν σε λαβεί σε αυτήν την περίπτωση. Δεν πρέπει να υποσκάψουμε τι καλέ σκέψεις μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένου Βασιλείου και Ινδίας, αλλά πιστεύω σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητο να κάνουμε κάποιε αιτήσει προ την κατεύθυνσή του. Οι Ινδοί μπορεί να έχουν πραγματικά ανησυχίε που είναι θεμητέ σε σχέση με παράνομη κατοχή όπλων και το κατανοώ αυτό μετά από τι επιθέσει στο Μουμπάι το 2008. Αλλά από ό,τι μπορώ να πω, οι Βρετανοί ε, οι Βρετανοί φρουροί, μεταξύ των οποίων και ένας από την εκλογική μου περιφέρεια, είχαν την λογική προσδοκία ότι δρούσαν σύμφωνα με τον νόμο, πιστεύανε ότι αγωνίζονται κατά της πειρατείας. Δούλευαν για μια αμερικανική εταιρεία. Δεν θεώρησαν ότι κάναν κάτι το οποίο να αντιβαίνει στο νόμο ή στα συμφέροντα της Ινδίας. Ούτε καν ξέρουν ότι τα όπλα τους τα είχαν παράνομα στην κατοχή τους. Αναρωτιέμαι λοιπόν κατά πόσο η συνεχιζόμενη φυλάξη τους εξυπηρετεί κάποιο συμφέρον. Καλό. Λοιπόν την ειδική κυβέρνηση να επανεξετάσει το θέμα αυτό και να απελευθερώσει τους Βρετανούς, Ιταλούς και Εστονούς πολίτες οι οποίοι βρέθηκαν σε καταστάσεις για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνοι. Ευχαριστώ. Διαδικασία Catch Ο Καπούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πέρασε ένας χρόνος από τότε που με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίναμε ένα ψηφίσμα για το θέμα των Ιταλών αυτών που συνελήφθησαν στην Ινδία το 2012 και που ο εφιάλτης τους δεν γνωρίζει τέρμα. Ε, μπροστά στο αυθαίρετο δικαστήριο αποφασίστηκε η υπόθεση του ψηφίσματος να μην εξεταστεί στην ε, δικαιοσύνη. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε αυτό αυτή την περίπτωση ως μια πράξη αδυναμίας της Ευρώπης. Πριν από λίγους μήνες επαναλάβαμε με σαφήνεια ότι η κράτηση των ε, ναυτών αυτών είναι μια κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι Ιταλοί ναύτες όπως και όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κρατώνται στην Ινδία θα πρέπει να προστατευτούν όπω τα θελημένα τα δικαιώματά του. Και καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση γι' αυτό. Μέσα σε όλη αυτή την αυθαιρεσία, η Ινδία θα πρέπει να γνωρίζει ότι ό,τι απόφαση και να λάβει, αυτό θα έχει αντίκτυπο στι σχέσει τη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Γιάκοφτσιτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζω ότι καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια και θέλετε και να μιλάτε ο καθένας, στον καθένα στη γλώσσα του. Μιλάτε ζάμινικο όμως για μας όταν απευθύνεστε. Σάστοπνικ είναι η λέξη που σημαίνει βουλευτής. Σάστοπνικ. Θα ήθελα όμως τώρα να περάσω στην ουσία και να επιστήσω την προσοχή σας σε μια παράλογη κατάσταση οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να, να προστατεύσουν αυτούς και ε, αλλήλους από την ε, πειρατεία. Και τελικά αυτοί μπήκαν φυλακοί. Τι έγινε τώρα. Κρατούνται οι άνθρωποι αυτοί και ίσως και να μείνουν στη φυλακή πέντε χρόνια. Αν δεν τους ε, σώσουμε με τη διπλωματική μας δράση. Να τονίσω το εξής. Είναι παραγωγή η απαλληφή ε, της αναφοράς στους Ιταλούς ναυτικούς. Υπόθηκε. Ε, ίσως πράγματι να ισχύει όμως αυτό γιατί τους βοηθούμε με άλλους τρόπους. Ευχαριστώ. Ε, ε, η κυρία Κριστίνα Μορβάη τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι μεταξύ των ε, ανήκω στους ευρωσκεπτικιστές. Είμαι όμως και ποινικολόγος. Και πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα κάθε φορά όταν βλέπω τις προσπάθειες που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσει οποιονδήποτε ε, έχει συλληφθεί σε μια τρίτη χώρα, παρέχοντας μεταξύ άλλων και προξενική προστασία. Βέβαια, οφείλω να πω κάτι προς τον κύριο Ντέβα. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Ντέβα ότι μπορούμε να κάνουμε μαθήματα στην Ινδία σε ό,τι αφορά τις ποινές κάθυρξης. Στην περιφέρειά μου έχω έναν άνθρωπο ο οποίος ε, κρατήθηκε σε προσωρινή κράτηση για τρεις μήνες στη Ρουμανία γιατί δεν προσπαθούν να βρουν κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο απέναντι του ρουμανικές αρχές και σε όλη τη διάρκεια αυτή τη κράτηση δεν έχει καμιά επαφή με του οικείου του. Ήδη δηλαδή τιμωρεί το άνθρωπο. Δέχεστε κυρία Μορβά ε, μπλε κάρτα. Uh, will Madam accept? Κυρία, κυρία Μορβάη, δέχεστε ότι τους σύγχρονους καιρούς το να παραμένουν στη φυλακή κάποιοι σε κάθεξη για δύο χρόνια χωρίς εκδίκαση της υπόθεσής τους είναι κάτι απαράδεκτο. Μόνο αυτό είπα ότι χρειάστηκαν δύο χρόνια ώστε οι ειδικές αρχές να εξετάσουν σε επίπεδο δικαστηρίου και να προβλέψουν κάποια απόφαση για τους ανθρώπους αυτούς δεν ε, είχαν ε, κάνει κάτι άλλο παρά να εκτελέσουν ε, διαταγές οι άνθρωποι αυτοί. Και αν δεν τις είχαν εκτελέσει θα είχαν εκτελεστεί οι ίδιοι. θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ανάλογη μεταχείριση και θα πρέπει να έχουν προσέλθει ενώπιον της δικαιοσύνης νωρίτερα. Συμφωνώ απολύτως κύριε Ντέβα. είναι απαράδεκτο να μένουν στη φυλακή προεξέταση της υπόθεσής τους προδικαστικά άνθρωποι αυτοί είναι υπεραρκετό το διάστημα για να οργανωθεί η εκδίκαση. Και συμφωνώ και με τα υπόλοιπα επιχειρήματά σας, όμως παρόμοια προβλήματα έχουμε και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωση. Και είναι εξίσου ανυπόφορο αυτό και εξίσου παράλογο. Και γι' αυτό κάτι θα έπρεπε να γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Μουρβάη, δέχεστε κι άλλη γαλάζια κάρτα από τον κύριο Φρουτζουλίτσα. Ε, dear colleague Morvai, you said that you are a... Κυρία Μορβάη, είπατε ότι είστε δικηγόρος ποινικών υποθέσεων και μιλάτε για έναν Ούγκρο που κρατείτε στην Ρουμανία. Ξέρετε με τι κατηγορίες γιατί έχει φυλακιστεί στη Ρουμανία ο Ούγγρος αυτός πολίτης και υπάρχει και συμφωνία Ρουμανίας-Ουγγαρίας ως ε, κατώ μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνεργασία σε τέτοια ζητήματα. Δεν έχει καμία σχέση με έναν πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης που κρατώνται στην Ινδία. Ή το παράδειγμά σας. Κοιτάξτε, είμαι... Ε, Απόλυτα ενσυνείδητη του γεγονότος ότι, ένας, ότι πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες <clears throat> κατηγορούνται ε, για πρόθεση διάπραξης τρομοκρατικών ενεργειών. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι εδώ και τρεις μήνες στη φυλακή <clears throat> και οι αρχές εκεί δεν έχουν καταφέρει να παρουσιάσουν κανένα στοιχείο εναντίον των, ε, του ατόμου αυτού. Οι ρουμανικές αρχές όσο σοβαρό και να είναι το θέμα αυτό, ένα άτομο το οποίο βρίσκεται στη φυλακή θα πρέπει να διατηρήσει την επαφή με την οικογένειά του γιατί η προφυλάξη δεν πρέπει να είναι τμήμα της ε, τιμωρίας του. Ο κύριος Μιμίκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμβολή σας στη συζήτηση αυτή που αφορά στο ψήφισμα που καταλήγει με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς συμμεριζόμαστε τι ανησυχίε πολλών από εσά δύο χρόνια αβεβαιότητας έχουν οδηγήσει σε μεγάλη αγωνία όλων των ενδιαφερομένων. Παρακολουθήσαμε από πολύ κοντά την κατάσταση των φυλάκων από την Εστονία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαστε σε επαφή με τις εστονικές και βρετανικές αρχές σε ό,τι αφορά την προστασία αυτών των πολιτών. Έχει αναφερθεί πολλές φορές το θέμα αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τους Ινδούς συνομιλητές μας τους τελευταίους μήνες έχει αρνητική επίπτωση στον παγκόσμιο αγώνα κατά της πειρατείας σε μια στιγμή που η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη συνεργασία για να αντιμετωπιστούν αυτές οι απειλές. Μάθαμε πρόσφατα ότι ένα δικαστήριο στην Ταμίλ Ναντού καταδίκασε τους φρουρούς αυτούς των πλοίων σε πενταετή ε, φυλάκιση ενώ το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τους είχε αθώσει. Ξέρουμε ότι τώρα θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα μία προσφυγή στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω όλα αυτά που είπε η κυρία Μαρίνα Καλιούραν, η Υπουργός Εξωτερικών της Εστονίας, ότι από ανθρώπινη άποψη εγώ ήλπιζα <clears throat> να υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα, ανεξάρτητα όμως από το αποτέλεσμα θα συνεχίσουμε να δρούμε για να μπορέσουν να γυρίσουν οι άνθρωποι αυτοί στο σπίτι τους. Πρέπει να βρεθεί μια λύση το ταχύτερο δυνατό. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας μαζί με τις αρχές της Εστονίας και του Ηνωμένου Βασιλείου τις επόμενες εβδομάδες στις επόμενες φάσεις της δικαστικής διαδικασίας. Για τους δύο Ιταλούς ναύτας. Σέβομαι ιδιαίτερα το περιεχόμενο του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο θα εγκριθεί σήμερα, θα ψηφιστεί σήμερα αλλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί το ταχύτερο μια λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει το θέμα αυτό τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε όλα τα επίπεδα με, την, με τις συνδικές αρχές, ζητώντας να υπάρξει ταχεία και συνενετική λύση επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου σημαίνει όχι μονάχα συμμόρφωση <clears throat> με, το, με, τη, με, την νομοθεσία για τη θάλασσα των Ηνωμένων Εθνών αλλά και με, την, το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να υπάρξει διεθνής διαιτησία στα θέματα της ούγκλος με τρόπο ο οποίος να είναι συμβατός με το διεθνές δίκαιο. Έντιμα μέλη. Μπορείτε να είστε πεπισμένοι ότι εμεί θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σε κράτηση στην Ινδία και να συντονίσουμε τις ενέργειές μας με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Έχω λάβει ένα σχέδιο ψηφίσματος το οποίο θα περατώ στη συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει μετά το τέλος της συζήτησης.